ευρωπαϊκή οικονομία. Thank you, Commissioner. The debate is now closed. Σας ευχαριστώ. Τώρα ολοκληρώνεται η συζήτηση και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Θα αλλάξουμε η Επίτροπη. Θα δώσουμε λίγο χρόνο στον Επίτροπο Ναύεσης για να ε, καθίσει. Θα το συνεχίσουμε. Το επόμενο θέμα είναι η κοινή συζήτηση για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των διεθνών ζευγαριών. Δύο εκθέσεις του κυρίου Καβαντά. Μία για το, τη δικαιοδοσία εφαρμοστεί για αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και η δεύτερη για θέματα ε, για τα ίδια θέματα στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων ε, καταχωρισμένων συντρόφων. Ο κύριος Καβαντά έχει το λόγο 4 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Έξι μου είχαν προαναγγείλει. Θα προσπαθήσω να τηρήσω τα τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η κινητικότητα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μια ψευδέσεις. είναι μια πραγματικότητα. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 16 εκατομμύρια πολυεθνικά ζευγάρια ή διεθνή ζευγάρια ε, και έχουν αυτοκίνητα, σπίτια ή τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορες χώρες και σε περίπτωση προβλήματος ε, είναι ε, πραγματικά γολγοθάς για να βρούνε πώς, το, ποιο είναι το εφαρμοστό δίκαιο, πώς θα εκτελεστούν οι αποφάσεις, πώς θα μοιραστούν τις ευθύνες. Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου θα εκλείψει με αυτή τη νέα πρόταση για αυτά ε, και μην ξεχνάμε και το κόστος που επιστρέφουν αυτές οι περίπλοκες διαδικασίες στα διαζύγια, το, ε, στα, στους δικαστικούς ε, χωρισμούς ή σε περίπτωση θανάτου. Ε, και σε συγκρούσεις ε, που προκύπτουν από αυτές ε, τις δίκες. Οι νέες διατάξεις ισχύουν για, τα, για συζύγους ή για τα καταχωρισμένους συντρόφους. Πρέπει να γνωρίζουν τα ζευγάρια αυτά ποια είναι η αναγνωρισμένη δικαιοδοσία για τα περιουσιακά του στοιχεία που ενδεχομένω βρίσκονται σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. υπάρχουν άλλες διαφορές στα εφαρμοστέα δίκαια ανάλογα με τις χώρες και οι σύζυγοι οι σύντροφοι βάσει τη νέα πρόταση υπό ορισμένε προποθέσει θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την αρμόδια ε, δικαιοδοτική αρχή ε, στη χώρα ε, διαμονή, παραδείγματο χάρη, ή στη χώρα όπου οι σύζυγοι οι σύντροφοι έχουν την υπηκότητά τους και θα είναι ιδιαίτερα ευέλικτη αυτή η διάταξη θα ισχύει για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ακόμη και αν βρίσκονται σε άλλες χώρες σε σχέση με τη χώρα διαμονής. Ε, τονίζω ότι θα ε, εφαρμοστεί το δίκαιο όλων των χωρών ε, και θα τηρείται η αρχή της επικουρικότητας, διότι αυτοί οι δύο νέοι κανονισμοί δεν σχετίζονται με τον ορισμό του, των γαμικών σχέσεων ή των σχέσεων ε, μιας ε, καταχωρημένης σχέσης, διότι διέπονται, εξακολουθούν να διέπονται αυτές οι σχέσεις από τα εθνικά δίκαια. Ε, όταν μια χώρα δεν αναγνωρίζει μια τέτοια σχέση θα έχει τη διακριτική ευκαιρία να μην επιληφθεί μια τέτοια ε, διαφοράς ε, που προκύπτει στη συγκεκριμένη χώρα σε περίπτωση διαζυγίου δικαστικού χωρισμού ή θανάτου του συζύγου ή συντρόφου και θα μπορέσει να αναπέμψει το ζήτημα στο δικαστήριο μιας άλλης χώρας που εκείνη αναγνωρίζει την καταχωρισμένη σχέση. Ε, ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, όπως το γνωρίζετε, η συμφωνία ως προς το οικογενειακό δίκαιο χρειάζονταν η ομοφωνία, οπότε ε, αυτή η κατάσταση που οδηγεί σε μαρτύριο για πολλούς ανθρώπους χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να λήξουμε σε συμφωνία. 18 κράτη-μέλη, με θυμίζω, δέχτηκαν να εφαρμόσουν ε, αυτές τις νέες διατάξεις ε, στις μεταξύ τους σχέσεις. στη τελευταία ολομέλεια τον Ιούνιο του 2016 έδωσε τη συγκατάθεσή του, τη σύμφωνη γνώμη του μάλλον του Κοινοβούλου για την ενισχυμένη συνεργασία για αυτούς τους δύο κανονισμούς ε, για τα κατοχωρισμένα ζευγάρια και για τις γαμικές σχέσεις ε, με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν ε, συνέτρεξε καμία μεγάλη δυσκολία. Υπάρχει μια καλοπιστική διάταξη που προβλέπει ότι ε, υπάρχουν κάποιες χώρες που ε, μελλοντικά θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτή την ενισχυμένη συνεργασία. Κατά τη γνώμη είναι λίγο περίτη αυτή η διάταξη. Τέλο πάντων, σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την ουσία αυτών των προτάσεων. Η ομάδα μου και ο φαινόμενο προτείνουμε να καταψηφίσετε αυτή την τροπολογία διότι θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να τεθεί εν κινδύνο αυτή η συμφωνία προϊόν δύσκολων διαπραγματεύσεων ε, και που επιτρέπει την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ μια σειρά χωρών. Ε, είναι πολύ σημαντική η ψηφοφορία αύριο, διότι υπάρχει το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι σημαντικό να τηρηθεί, ούτω ώστε το Συμβούλιο τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτή την ενισχυμένη συνεργασία να μπορέσουν να εγκρίνουν αμελητή ε, τη νέα πρόταση. Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, μην ξεχνάτε πως πρόκειται για ένα συγκεκριμένο μεγάλο αριθμό ζευγαριών, 16 εκατομμύρια, 32 εκατομμύρια ανθρώπων, ε, καταλαβαίνετε πόσες ε, οικογένειες ε, εμπλέκονται και θα διευκολυνθεί η ζωή τους με αυτές τις αποφάσεις. Ευχαριστούμε, Επίτροπος Ναυραζίτης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. <clears throat> Αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Οι Ευρωπαίοι πολίτες κάνουν χρήση του δικαιώματός τους ελεύθερης διακίνησης και κατάστασης. Σήμερα υπολογίζονται σε 16 εκατομμύρια τα διεθνή ζευγάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συχνά αντιμετωπίζουν τις χέρειες στη διαχείριση της περιουσίας τους ή σε περίπτωση θανάτου ή διαζυγίου, όταν πρέπει να χωριστεί η περιουσία. Οι νέοι αυτοί κανόνες, σε ό,τι αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας διεθνών ζευγαριών, ε, έγκαμων ζευγαριών αλλά και καταχωρισμένων σχέσεων, έχουν στόχο <clears throat> να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσχερίες... και να προσφέρουν σε διεθνείς οικογένειες ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά και τις διαδικασίες όταν τα πράγματα πάνε άσχημα. Θα γνωρίζουν τα ζευγάρια με σαφήνεια ποιο είναι το κόστος που συνεπάγεται ο χωρισμός της ε, κυριότητας και τι μέτρα θα πρέπει να λάβουν. Νέοι κανόνες λοιπόν που βασίζονται και σε αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων σε εμπορικά και ε, πολιτικά θέματα, όπως έχει εγκρίνει το Συμβούλιο ήδη ε, πριν από ένα χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή σας, κύριο Καβαντά, για την συνεργασία στην προώθηση του σημαντικού και δύσκολου αυτού θέματος. Σε ενισχυμένη συνεργασία. Θα θέλαμε βέβαια τα σημαντικά αυτά θέματα να είχαν λυθεί με συμμετοχή όλων των χώρων μελών. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε τώρα, βασιζόμενοι στις χώρες μέλη που επιθυμούν και να δεχθούμε και τις άλλες χώρες όταν αυτές θα θεωρήσουν ότι μπορούν και πρέπει να συμμετάσχουν. Στο μεταξύ, οι κανόνες της ενισχυμένης συνεργασίας περιλαμβάνουν και διατάξεις για τις ρυθμίσεις για τα ε, διεθνή ζευγάρια, και στην ενισχυμένη συνεργασία και οι χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν για χώρες μάλλον όπου, που δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία δεν θα ισχύουν οι κανόνες αυτοί. Επιθυμώ να διαβεβαιώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι τα σχέδια κανονισμών περιλαμβάνουν και διασφαλίσεις για, την πλήρη, για τον πλήρη σεβασμό των νομικών παραδόσεων των χωρών μελών. Δεν εμπλέκονται στην αναγνώριση καταχωρισμένων ζευγαριών σε άλλε χώρε μέλη. Θα ισχύσουν οι κανόνε αυτοί, ελπίζω, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο κύριο Βόση για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνω πρώτα τι ευχαριστίες μου και εγώ στον εισηγητή, αλλά και στην προκάτοχό μου που χειρίστηκαν πάρα πολύ καλά το θέμα είναι απίστευτο ότι μόλις τώρα ερχόμαστε να εγκύψουμε σε τέτοια θέματα και νομοθετικά δηλαδή διότι βεβαίως έχουμε την ελευθερία διακίνησης εδώ και τόσες δεκαετίες. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα ένιωθαν ε, μοναξιά αν έβλεπαν πώς πόσο περίπλοκες είναι οι διαδικασίε που βλέπει το ιδιωτικό διεθνέ δίκαιο για τον χωρισμό περιουσιών, για παράδειγμα, σε ε, περιπτώσει όπω προαναφέρθηκαν. Και η ψηφοφορία αύριο για την ενισχυμένη συνεργασία ορισμένων χωρών μελών στα θέματα αυτά του εμπράγματου δικαίου και για γάμου αλλά και για καταχωρισμένα ζευγάρια αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στο τέλο πολιετών διαπραγματεύσεων. Χρειαζόμαστε επιγόντω τι ρυθμίσει αυτέ και είναι μεγάλο το ενδιαφέρον μας ως συνομοθέτου να ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέματος αυτού εδώ στην Ολομέλεια. Βρισκόμαστε στη διαδικασία της ακροάσεως, θα έλεγα, ακόμα. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα για το γεγονό ότι το Συμβούλιο δέχτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό όλες τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την πορεία Τη υποθέσεως ως τώρα. Και βεβαίως τα κείμενα έχουν γίνει ε, δεκτά και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ευτυχώς φροντίσαμε και για το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν ένομες συνέπειες σε ό,τι αφορά την αναγνώριση μορφών συμβιώσεως που ακόμα δεν γνωρίζουν στην νομοθεσία τους ορισμένες χώρες μέλη. Διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε ενδεχομένω σε παραπέρα μπλοκαρίσματα. Είναι καλό λοιπόν που το κείμενο περιλαμβάνει και ρήτρα δημοσία τάξεω για τα αναγνωρισμένα ζευγάρια. Βρίσκω ότι η λύση αυτή που δόθηκε είναι πιο σωστή. Και ε, συγχαίρω και ευχαριστώ όλε και όλου όσοι συμμετέσχουν. Ευχαριστώ. Για τρία λεπτά η κυρία Κέπχαρτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που επιτέλους σήμερα φτάνουμε στην ολοκλήρωση της συζητήσεως αυτής στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία είχα αναλάβει τότε την ε, έκθεση. Ήμουν εισηγήτρια δηλαδή. Και τώρα ήμουν συνεισηγήτρια. Μακρά διαδικασία για να δώσουμε λύσεις στους πολίτες και των δύο φίλων δηλαδή διεθνών ζευγαριών για να μπορέσουν να απολαύσουν τις ελευθερίες που τους εξασφαλίζουν οι συνθήκες και σε ό,τι αφορά την γονική μέρημνα και σε ό,τι αφορά τώρα πλέον και το εμπράγματο δίκαιο, θεωρώ ότι κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Δηλαδή δίνουμε μια χείρα βοηθείας στους ανθρώπους εκείνους που είπαν θα την ζήσουμε αυτή την Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη σε όλη τη τη διεθνική διάστηση. Είναι καλή, καλό πράγμα αυτό λοιπόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρχή θεώρησε ότι είναι πολύ σημαντικό να φροντίσει ότι οι δύο νομοθετικές προτάσεις που έχουν τεθεί επιτάπητος, δηλαδή αφενός για τα καταχωρισμένα ζευγάρια και αφετέρου για τους γάμους, ότι και οι δύο αυτές ε, ρυθμίσεις δηλαδή περιλαμβάνουν κατά βάση τα ίδια δικαιώματα. Ταυτόχρονα όμως σέβονται τις διαφορετικές παραδόσεις και τον διαφορετικό νομικό πολιτισμό των διαφόρων χωρών μελών. Γι' αυτό ειδικά αυτή η ρήτρα που λέει ότι καμία χώρα μέλος δεν πρόκειται να εξαναγκαστεί να θεσπίσει τον θεσμό των αναγνωρισμένων ζευγαριών, εφόσον δεν τον έχει στην νομοθεσία τη ή δεν τον επιθυμεί. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ρήτρα. Σημαντικό επίση στα πλαίσια του νομοθετήματο αυτού ήταν για μα, του σοσιαλδημοκράτε, να πούμε ότι δεν θα υπάρξει άγρα δικαστηρίου, forum shopping. Τα είδαμε αυτά. Είδαμε δηλαδή ότι ο ισχυρότερο ή ο πλουσιότερος των δύο εταίρων, των δύο συντρόφων, όταν ετίθεται το θέμα χωρισμού ή διαζυγίου, επέβαλε την βούλησή του και οδηγούσε τον ασθενέστερο σε μειονεκτική θέση. Νομίζω ότι μπορέσαμε με τη ρύθμιση αυτή να το αποφύγουμε. Μπορέσαμε να φτιάξουμε ένα δίκαιο λοιπόν όπου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβουλίο των Υπουργών δέχτηκαν τελικά και ακολούθησαν τι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό να μας ακούσουν, διότι εν τέλει μπορέσαμε να συναποφασίσουμε το περιεχόμενο των νομοθετημάτων. Με αυτή τη δουλειά μας λοιπόν θεωρώ ότι μπορέσαμε να φροντίσουμε για άλλη μια φορά να λύσουμε πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων που τα ζουν καθημερινά. Ευχαριστώ πολύ και για ένα λεπτό ο κύριος Τζαμπάσκι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Το οικογενειακό δίκαιο είναι πολύ λεπτό θέμα και θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να το προσεγγίσουμε. Πρόκειται για ένα τομέα που ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο εν γέννη. Τα τελευταία χρόνια είχαμε αυξημένη συνεργασία σε πολλούς νομικούς τομείς ένας εξ αυτούς είναι ο τομέας των διασυνοριακών νομικών ε, δράσεων. Όμως οι εθνικές ε, διατάξεις συχνά διαφέρουν εδώ. Για παράδειγμα, όταν αφορά τις ε, καταχωρημένες σχέσεις, αυτό δεν ισχύει στην Ιταλία, την, Πολωνία, την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Ε, επίσης, είναι αντιφατικά ζητήματα μπορεί να δημιουργηθεί έτσι νομική αβεβαιότητα. Και θα ήθελα να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να προσέξουμε εδώ εγώ είμαι υπέρ της καλύτερης συνεργασίας, ωστόσο πρέπει να επιμείνουμε στην αρχή της αναλογικότητας. Ο κύριος Χρυσόχωνος τώρα. Δίνουμε σήμερα την έγκρισή μας για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στους τομείς της διεθνούς δικαιοδοσίας του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων στα ζητήματα περιουσιακών σχέσεων συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων. Οι νέοι κανόνες μεταξύ των 18 κρατών μελών που συμφώνησαν να συμμετάσχουν στο καθεστώς ενισχυμένης συνεργασίας αναμένεται να διευκολύνουν την καθημερινή ζωή ζευγαριών υπηκών διαφορετικών κρατών μελών με την επιλογή ενός νομοθετικού πλαισίου που θα εφαρμόζεται στα περιουσιακά του στοιχεία καθώς και με την καθιέρωση της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων που εκδίδονται σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Είναι πραγματικά λυπηρό ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής το 2011 δεν προχώρησε λόγω έλλειψης ομοφωνίας στο Συμβούλιο με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστερήσει πέντε χρόνια να θεσπίσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες. Επίσης λυπηρό είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει απλώς τη γνώμη του στα ζητήματα οικογενειακού δικαίου, όπως αυτό που συζητούμε σήμερα, και που έχει άμεσες επιπτώσεις σε χιλιάδες ζευγάρια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για ανάλογα ζητήματα θα έπρεπε να εμπίπτουν στον τομέα της συναπόφασης, ώστε να μπορεί το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ως ο άμεσος εκπρόσωπος των ευρωπαίων πολιτών να έχει λόγο σαν ισότιμος εταίρος στην νομοθετική διαδικασία και να επηρεάζει αποφασιστικά τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. λεπτά, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πώς μπορούμε να ανεχόμαστε μια κατάσταση όπου μια οικογένεια, οι γονείς με τα αγαπημένα τους παιδιά ή ε, ένα ζευγάρι που έχει υποσχεθεί, έχουν υποσχεθεί ε, αιώνια ζωή να χάσουν το δικαίωμά του αν μετακινηθούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Πώς μπορούμε να ανεχόμαστε μια κατάσταση όπου οι γονείς δεν μπορούν να κάθονται Δηλαδή κοντά στα παιδιά τους στο νοσοκομείο αν έχουν ένα ε, ατύχημα επειδή είναι πέρα από τα σύνορα. Και πώς μπορεί μια οικογένεια να χάνει τα διεκτησιακά της δικαιώματα επειδή κάποια κράτη-μέλη δεν καταλαβαίνουν ότι η οικογένεια και ζευγάρι και η αγάπη ε, μπορεί να πάρουν διάφορες μορφές. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν και πιστεύω πως αυτή η πρόταση είναι ένα μικροσκοπικό πρώτο βήμα για αυτή την, προς αυτή την κατεύθυνση οι, οι οικογένειες ίδιου φύλου δεν μπορούν, τα, τα, τα ζευγάρια ίδιου δεν μπορούν να είναι δεύτερη κατηγορία πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται να μπορούν να λένε ελεύθεροι να κινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εργάζονται, να σπουδάζουν όπου θέλουν και να προστατεύονται από τι διακρίσει. Αυτό δεν είναι κάτι το υπερβολικό. Ένα δικαίωμα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ας, ε, πάψει πάψουν οι διακρίσεις κατά των ζευγαριών ίδιου φύλου ε, και το, κατά των οικογενειών του ουρανίου τόξου. Α ε, φτιάξουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει στήριξη και προστασία σε όλε τι οικογένειε. Αυτή η πρόταση είναι ένα μικρό κομμάτι ενό μεγάλου παζλ ώστε να γίνει αυτό πραγματικότητα. Α το πάρουμε αυτό σημείο κίνηση για να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου όλε οι οικογένειε και όλα τα ζευγάρια να μπορούν να ζουν όπω επιθυμούν και να κινούνται όπω θέλουν και να έχουν τα ίδια δικαιώματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά, Φαν Στόρχ. Ευχαριστώ. Μιλούμε για δύο νομοθετήματα τα οποία περιλαμβάνουν και τον ορισμό της οικογένειας. Ήδη προετών το Συμβούλιο Υπουργών είχε καταθέσει ρύθμιση για τη ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων των ζευγαριών. Τώρα για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Η Πολωνία τον μπλοκάρισε διότι δεν γνωρίζει το θεσμό αυτό. Πρόκειται όμως για προσέγγιση γραφειοκρατική. Πάνε λοιπόν με αυτά τα πράγματα να βάλουν την, τον γάμο ομοφιλοφίλων από την πίσω πόρτα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωμη ε, Τάξη. Υποσκάπτοντας έτσι τις εθνικές συνταγματικέ διατάξεις. Αυτές είναι οι ιδέες Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρίπτουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση γεννώνται ιδέες που υποτίθεται ότι πρέπει να τις αποδεχτούν εν τέλει όλοι. Και αν δεν τους αποδεχτούν, τους βρίζουν και τα βάζουν μετά από την πίσω πόρτα. Γι' αυτό και υπάρχει μια πανευρωπαϊκή υπάρχει μια πανευρωπαϊκή κίνηση που επιγράφεται πατέρας, μητέρα, παιδιά και που έχει ως σκοπό να γίνεται δεκτός ο γάμος μόνο ως γάμος. Ο γάμος αποτελείται από γυναίκα και άνδρα. Έναν άνδρα και μια γυναίκα. Τελεία. Πάψτε να τα θεωρείτε αυτά διάκριση. Ούτε να τα χαρακτηρίζετε ως κάτι το άρρωστο, ως φοβία. Ο γάμος είναι κάτι διαφορετικό από ένα αναγνωρισμένο, ένα καταχωρισμένο ζευγάρι. Δεν είναι τίποτα καλύτερο ή χειρότερο, είναι απλώς διαφορετικό. Όσοι θέλουν να κρατήσουν αυτό το θεσμό της οικογένειας, λέω επαγρυπνείτε. Από τούτην εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορείτε να περιμένετε τίποτα καλό. Είναι μεν ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι πολίτες είναι ισχυρότεροι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σύμφωνα με την Κομισιόν των Βρυξελών υπάρχουν 16 εκατομμύρια διεθνή ζευγάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι και αν ισχύει στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το παίρνει ως πρόσχημα για να ε, ε, ε, αναμειχθεί στα, δικ, στα στο οικογενειακό δίκαιο. Το ένα αφορά να αναγνώριση των γαμικών καθεστώτων. Θα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη να κυρώσουν τη συμφωνία που υπάρχει εδώ και χρόνια. Επίσης, δεύτερη ανάμεξη σε όλα αυτά είναι το θέμα της αναγνώρισης των ε, καταχωρημένων σχέσεων. Και εδώ υπτίθεται πρόβλημα γιατί κάθε κράτος έχει τη δική του αντίληψη. Το να θέλουμε να επιβάλλουμε την αναγνώριση ξένων ε, καταχωρημένων σχέσεων θα αντιστοιχίσει στην ε, παράκαμψη των εθνικών κανόνων σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό 10 κράτη από τα 28 αρνήθηκαν να δεχτούν αυτά τα δύο κείμενα και γι' αυτό και εγώ θα τα καταψηφίσω. Σας ευχαριστώ. Και τώρα για δύο λεπτά, Εσταράς Φεραγκούτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως συζητάμε ένα θέμα που έχει ιδιαίτερη σημασία και θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία ε, στον κύριο Καβαντά ε, τον εισηγητή. Υπάρχουν διάφορες πρακτικές και νομικές δυσκολίες ε, και για λόγω, ε, γιατί υπάρχουν διαφορετικέ νομοθεσίε που ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση. Είτε πρόκειται για γάμο, είτε πρόκειται για διαζύγιο. Γι' αυτό και έπρεπε να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση όσον αφορά αυτέ τις καταχωρημένε ε, σχέσεις και να τα αντιμετωπίσει η Ένωση αυτό το θέμα. Δεν υπήρξε ομοφωνία και γι' αυτό και τα 17 κράτη-μέλη ζητάνε ενισχυμένη συνεργασία για να, βοηθήσουν, να, να διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών. Θέλουμε να αποσαφηνίσουμε νομικό στο θέμα, να, να ορίσουμε ποιο έχει αρμοδιότητα, ποιο είναι το αρμόδιο ε, νομικό όργανο, ποιο είναι το ε, εφαρμοστέο δίκαιο και επίσης ε, να εφαρμοστούν όλες αυτές τα ψηφίσματα γιατί η ελεύθερη κυκλοφορία είναι μία από τις προτεραιότητες της Ένωσης η διαδικασία θα πρέπει να είναι πολύ πιο γρήγορη και πιο ασφαλής. Αναμφίβολα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρά τα διαφορετικά νομικά συστήματα των ευρωπαϊκών κρατών. Και επίση έτσι θα τεθεί τέλο σε διάφορε συγχύσεις και μπερδέματα. Αυτό το πράγμα είναι θελοντικό. Όποιο κράτο μέλο θέλει θα μπορεί να προσχωρήσει και θέλουμε να δυσκολύνουμε τη ζωή των πολιτών της Ένωσης. Στην πράξη πρόκειται για ένα ε, μέσο ε, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που έρχεται να συμπληρώσει τα πολλά και διάφορα μέσα που υπάρχουν ε, στο αστικό δίκαιο και στο οικογενειακό δίκαιο συγκεκριμένα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα γιατί έτσι μπορούμε με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσουμε την αρχή της μη διάκρισης. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, σε ευχαριστώ. Επόμενος ο μας δεν είναι εντός αιθούσης, οπότε θα περάσω στον κύριο Σκρίπεκ. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι σημαντικός ο νομοθετικός αυτός στόχος και ένα σημαντικό μήνυμα. Γάμος, παιδιά. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Και για αυτά θέλουμε να υποστηρίξουμε εμείς ε, ευρωβουλευτές, τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρόκειται για αρνητική εξέλιξη ωστόσο αυτή η υπόθεση των καταχωρισμένων ζευγαριών. Εγώ τα θεωρώ αυτά καταστροφικά ως τάσεις. Οι πολίτες θεωρούν ότι του εξαπατούμε. Το ίδιο ισχύει και με την κύρωση της ε, Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Εάν το δεχθεί συνολικά αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα σημάνει άλλο ένα πλήγμα στην εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Εμείς είμαστε υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ των προέδρων στις καρέκλες τους. Sorry, you have a blue card. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, έχετε μια γαλάζια κάρτα. Δέχεστε. Έχετε 30 δευτερόλεπτα, κυρία. Κύριε Πρόεδρε, λέτε ότι τα δικαιώματα αυτά δεν θα πρέπει να καλυφθούν από ευρωπαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις. Μα κάθε χώρα μέλος έχει το δικαίωμα να το πράξει αυτό. Και ο καθένας έχει τα ανθρώπινα δικαιώματα του. Και όμως εσείς τα αρνείστε. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό είναι ικανοποιητικό. Πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Κυρία συνάδελφε, θα γνωρίζετε, θα γνωρίζετε κυρία συνάδελφε, ότι Ιδίω ε, συγκεκριμένα ο τομέας αυτός υπάγεται στην αρχή της επικουρικότητα Κάθε χώρα μέλο και η δική μου επομένω κρίνει και αποφασίζει μόνη της για τον τομέα αυτό. Όλοι έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα δικαιώματα. Κύριε Σφόβοντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κύριο Καβαντά για την εργασία του και για τις δύο αυτές προτάσεις. Ενισχυμένη συνεργασία, αυτό εμένα μου φαίνεται χρήσιμο πράγμα. Ήδη το 2007 είχε κάνει σχετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε βρει 13% των, διεθ... των γάμων να είναι διεθνείς. Είναι σωστό λοιπόν να δοθούν τα δικαιώματα αυτά διαμεθοριακά στα ζευγάρια αυτά και με τις νέες ρυθμίσεις θα υπάρξει εξοικονόμηση 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι δικαστικές δαπάνες που καλούνται να υποστούν τα ζευγάρια αυτά για να μπορέσουν να κάνουν δίκες σε διάφορες χώρες. Ο σκοπός, ωστόσο, του κανονισμού δεν είναι να εναρμονίσει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των διεθνών ζευγαριών. Οι προτάσεις που έχουμε μπροστά μας δεν λέγουν άλλωστε ότι τα καταχωρισμένα ζευγάρια εξισούνται με τα έγκαμα. Ο στόχος είναι να υπάρξουν ενοποιημένοι κανόνες για την διαίρεση της περιουσίας. Ε, βρίσκεται δηλαδή σε απόλυτη αρμονία με την αρχή της επικουρικότητας. Άλλωστε υπάρχει και η ρήτρα δημοσίας τάξεως που επιτρέπει σε κάθε χώρα μέλος που επιθυμεί να μην τον εφαρμόσει εφόσον υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που τις το επιβάλλουν. Εάν για παράδειγμα υπάρχουν διαφορές σε ό,τι αφορά τον ορισμό των καταχωρισμένων σχέσεων. Η ελευθερία διακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεμελιώδης. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη μεριά έχουμε και υποχρέωση να μην περιπλέκουμε την άσκηση αυτής της ελευθερίας Αντίθετα, να δημιουργήσουμε ένα κοινό χώρο με κοινού κανόνε διαμεθοριακά, όπω αυτοί οι κανόνε που συζητούμε σήμερα. 1,5 λεπτό, Γκασπάρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τον συνάδελφο Καβαντά για την εργασία του και για τη συνένεση που κατάφερε να φέρει στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων σε αυτό το θέμα. Ο κανονισμός αυτός ε, ε, οδηγεί σε ένα βήμα μπροστά, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, για όσον αφορά τα πραγματικά ε, δικαιώματα. Αυτός ο κανονισμός δίνει μια αναπάντηση συγκεκριμένη και βεβαιότητα νομική όσον αφορά αλλά και απλούστευση για τα 16 εκατομμύρια διεθνών ζευγαριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι πιο εύκολο να γνωρίζει κανείς την νομοθεσία, να εφαρμόσει την να ξέρει ποια είναι η δικαιοδοσία και ποια είναι η νομοθεσία που ισχύει. Μετά από την έναρξη ισχύω του κανονισμού στα 18 κράτη που στήριξαν αυτή την ενισχυμένη συνεργασία, θα μπορούν θα να προσταθούν κι άλλοι, έτσι ώστε να καταστεί ακόμα πιο αποτελεσματικό και συνεκτικός ο Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Ευχαριστώ τέλο την ε, Ολλανδική ε, Προεδρία που μπόρεσε να κλείσει θετικά αυτή τη διαπραγμάτευση και καλό και την ε, μελλοντική Σλοβακική Προεδρία να εργαστεί ώστε να επεκταθεί η συνένεση στο σύνολο των χωρών για αυτή τη μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά η κυρία Κομοντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόλι Μόλις στην τελευταία ολομέλεια το Κοινοβούλιο υπερψήφισε την μείωση της γραφειοκρατίας για τους Ευρωπαίους πολίτες, ιδιαίτερα κατά την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης. Όταν, ψηφίσαμε για την αναγνώριση των δημοσίων εγγράφων, αύριο με την κοινοβουλευτική ψηφοφορία θα υπερψηφίσω την έκθεση του κ. Καβαντά, έτσι ώστε τα διεθνή ζευγάρια στην Ένωση να έχουν ένα σαφές πλαίσιο ώστε να διαχειρίζονται την περιουσία τους. Σήμερα τα διεθνή ζευγάρια πιο ευάλωτες στιγμές ε, της ζωής τους είτε διότι διαλύεται ο γάμος τους ή η καταχωρημένη σχέση έχουν από πάνω να αντιμετωπίσουν και ένα σωρό δυσκολίες για το ποιο δικαστήριο θα είναι αρμόδιο και ποια νομοθεσία θα ισχύει. Συχνά μετά από ένα διαζύγιο, ένα χωρισμό ε, το, το ζευγάρι πρέπει να ξεκινήσει χωριστές διαδικασίες σε μια άλλη δικαιοδοσία ώστε να λυθούν ζητήματα που, που σχετίζονται με το καθεστώς ιδιοκτησίας. Αυτές οι δύο μεταρρυθμίσεις για την ενισχυμένη συνεργασία θα εξασφαλίσουν τη σαφήνεια και τη βεβαιότητα. Τα ζευγάρια θα έχουν να ακολουθήσουν απλοποιημένες διαδικασίες οπότε αν υπάρξει ζύγιο χωρισμός ε, θα είναι τα ίδια τα δικαστήρια που θα αποφασίζουν ε, ε, πιο καθεστώς ισχύει, δεν χρειάζεται να κάνουν και άλλες διαδικασίες σε καραταγμέλ και να μπλέκουν σε περίπλοκα νομικά ζητήματα για να βρουν το δίκαιο τους. Ε, ε, θα πρέπει θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για αποζημιώσεις και για, και για αποκατάσταση δικαστική. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Νεκρέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τις καταχωρισμένες σχέσεις και για τους γάμους οι ρυθμίσεις δηλαδή που ήρθαν τώρα είναι κάτι που έπρεπε να είχε γίνει πριν από πολύ καιρό. Πάλι καλά όμως έχουμε την πρόταση αυτή. Πρόκειται για προϊόν ενισχυμένης συνεργασίας και για κάποιες τροποποιήσεις. Ωστόσο, ο κανονισμός θα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για 16 εκατομμύρια διεθνή ζευγάρια που θα ε, ρυθμίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για τα θέματα αυτά. Ένα δίκαιο το οποίο πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις χώρες μέλη, έτσι ώστε να ισχύουν τα ίδια δικαιώματα για όλα τα ζευγάρια αυτά σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται ευκρινέστερη κατάσταση για τα ζευγάρια αυτά. Ευχαριστώ. Σέινφελτ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα ε, είναι προς συζήτηση ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σύγκριση με ένα ε, πολύ σημαντικό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το δημοψήφισμα για το Brexit. Δεν ξέρω αν είναι σημαντικό να το αναφέρω, θα δούμε σε ποια, κατεύθυνση θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μέλη γενέστε με, την, με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της. Είναι ανθρωπιστικού χαρακτήρα αυτή η Ένωση και ε, τα θεμέλια αυτής της Ένωσης ε, είναι η αρχή της ε, ανεκτικότητας. Τι θα γίνει ε, στο μέλλον, ποια πραγματικότητα θα ζήσουμε στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επίσης, συζητάμε ε, για το θέμα μιας δίκης που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, μιας ε, διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια και ολοκληρώνεται τώρα. στον ε, δημόσιο και στον ιδιωτικό βίο θα πρέπει να περιορίζουμε το κόστος και τα βάσανα που επισύρει μια τέτοια μακρόχρονη διαδικασία. Ελπίζουμε αύριο να ληφθούν οι ακατάλληλες αποφάσεις ούτως ώστε να διευκρινίσουμε ε, τις σχέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις σχέσεις ε, των πολιτών μεταξύ τους, τις σχέσεις που επικρατούν στην ευρωπαϊκή ε, κοινωνία για να είναι στο κέντρο αυτών των σχέσεων οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εξυπηρετούν τους πολίτες οι αρχές και θα ήθελα να να προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες και θα ήθελα αυτή την έκκληση ακριβώς ε, να απευθύνω. Θα πρέπει να υπομιστούμε τις ευθύνες μας ενώπιον των πολιτών. Ευχαριστούμε κυρία Ροντρίγκε. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε 13% ε, των ζευγαριών ε, βάσει των στοιχείων του 2017 ε, θα υποφεληθούν από αυτές τις νέες διατάξεις. Εάν προσθέσουμε στους γάμους και στους γάμους τα διαζύγια θα συνειδητοποιήσουμε ποιο θα ήταν το συμφέρον αν θα ήταν ήδη ξεκάθαρες οι διατάξεις για τις περιουσιακές σχέσεις των ζευγαριών. Βλέπουμε λοιπόν ότι για τις γαμικές διαφορές δεν επιλύεται το βασικό πρόβλημα αυτών των σχέσεων. Ε, Βεβαίω, το σημαντικότερο μέσο είναι ε, ε, οι περιουσιακέ σχέσεις των ζευγαριών ή των καταχωρισμένων συντρόφων, ώστε να μπορέσουν οι δικαστικές αποφάσεις να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναγνωρίζονται και να εκτελούνται ελεύθερα αυτές οι αποφάσεις στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπάμαι όμως που η δικαιοσύνη δεν επικράτησε στο Συμβουλίο, δεν υπήρξε η ομοφωνία, παρότι ήταν ευκαιρία. Θεό και αναγκαστήκαμε να ε, προσφύγουμε στην ενισχυμένη συνεργασία. Μόνο 18 ε, κράτη-μέλη αποφάσισαν ε, να έχουν εμπιστοσύνη το ένα στο άλλο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πόσπης. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, υποστηρίζω αυτές τις προτάσεις, όπως ακριβώς και οι συνάδελφοί μου. από την ομάδα μου. Έχουν περάσει 6-7 χρόνια από την αρχή των συζητήσεων στο Συμβούλιο. Εγώ ήμουν υπουργό δικαιοσύνη ε, τότε και συμμετείχαν στις συζητήσεις και προμηνιόντουσαν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Ε, ήλπιζα βεβαίως ότι θα επικρατήσει ο κοινός νους, ε, η κοινή λογική και ελπίζω το ίδιο να ισχύσει και αύριο και να εγκριθεί η πρόταση. Βεβαίως θα ισχύσει μόνο για 18 κράτη-μέλη και όχι ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα περιοριστούν οι οι ευνοϊκέ υποφελεί αυτέ τι διατάξει σε ένα μέρο των πολιτών. Σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται η κυριαρχία των κρατών μελών. Σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζονται οι αρχέ του οικογενειακού δικαίου των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και τίθεται το ζήτημα για τι καταχωρισμένε σχέσει αν ε, αναγνωρίζονται ή όχι από όλα τα κράτη-μέλη. τι πράγμα μιλάμε τελικά. Μιλάμε για ιδιωτικό δίκαιο ε, οικογενειακό δίκαιο για διοικονομικό ε, δίκαιο. Ένα θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο και επειδή είμαι από τον κλάδο ξέρω πόσο επωφελείς θα είναι οι διατάξεις. Ε, είχα πολλούς πελάτες ε, που διεθνεί ζευγάρια που είχαν πάρα πολλά προβλήματα διότι τα περιουσιακά τους ε, στοιχεία υπάγονταν σε πολλά διαφορετικά, πολύ διαφορετικά νομικά συστήματα. Δεν μπορεί κάποιος να αντιτάσσεται σε μια διάταξη που είναι επωφελής ε, για τους πολίτες. Δεν πρόκειται για περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας από πλευρά των Βρυξέλλων. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα υποστηρίξω την πρόταση παρότι λυπάμαι που δεν θα ισχύσει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα λεπτό κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η διαχείριση και η εκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων των διεθνών ζευγαριών λόγω χωρισμού του ζεύγου ή θανάτου ενό εκ των συζύγων εμπίπτει αρχικά στην αποκλειστική εθνική δικαιοδοσία. όμω το συμβούλιο προτείνει την αλλαγή αυτή τη κατάσταση θέλει να δημιουργήσει ένα ενιαίο καθεστώ ώστε το ζήτημα των περιουσιακών στοιχείων των διεθνών ζευγαριών να υπάγονται σε ένα διεθνέ δίκαιο. Όμως έτσι ο υποψήφιος κανονισμός ακυρώνει τα εθνικά δίκαια. Ακυρώνει τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που ισχύουν μέχρι σήμερα σε όλα τα κράτη-μέλη και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και στο τέλος οδηγεί στη δημιουργία ενός διεθνούς δικαίου η ρήτρα δημόσια τάξη αντιμετωπίζει με το πρόβλημα που έχει σχέση με την μη αναγνώριση σε ορισμένε χώρε ορισμένων σχέσεων συμβίωση δεν θεωρώ όμω ότι επιλύει τα νέα προβλήματα που δημιουργεί ο νέο κανονισμό αφού παραβιάζει την αρχή τη επικουρικότητα και δεν σέβεται τι πολιτισμικέ παραδόσει των κρατών μελών τη ένωση. επομένω θεωρώ ότι ο κανονισμό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει. ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλά νέα μου φαίνεται ότι είναι αυτά για 16 εκατομμύρια ζευγάρια Ευρωπαίων πολιτών που θα διευκολυνθεί η ζωή τους. Οι συζητήσεις διήρκεσαν για υπερβολικά μεγάλο διάστημα. Οι συζητήσεις για καταχωρισμένες σχέσεις, και για διεθνή ζευγάρια. Είναι απαράδεκτο που 10 χώρες μέλη δεν δέχονται την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του εισηγητού μας κύριου Καβαντά. Η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους είναι το ρότερο πράγμα στον κόσμο. Όμως, στην, ε, πάνω στην πραγματική ζωή, βεβαίως υπάρχουν και διαζύγια, υπάρχουν και ατυχήματα, υπάρχουν θάνατοι. Χρειάζονται τα διεθνή ζευγάρια ασφάλεια δικαίου. Αν δεν τα έχουμε αυτά, τι είδου αξίε θα χρησιμοποιήσουμε για να θεμελιώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Καπούτο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αυξανόμενη κινητικότητα των ανθρώπων σε ένα χώρο άνευ εσωτερικών συνόρων έχει οδηγήσει σε στη δημιουργία πολλών διεθνών ζευγαριών. 16 εκατομμύρια ε, ζευγάρια έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και σε περίπτωση διαζυγίου, χωρισμού ή θανάτου του εταίρου. Πρόκειται για το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο, τα θέματα ε, του γάμου λοιπά. Οπότε θα πρέπει να μπορούν όντως να διαλέξουν ε, το δίκαιο, να γνωρίζουν τι ισχύει, να ξέρουν την κυριότητα και την αναγνώριση του Ένωσης και τα λοιπά. Μεγάλο βήμα μπροστά είναι η αρχή της ενότητας ε, του εφαρμοστέου δικαίου που προβλέπει ότι τα γαμικά δικαιώματα θα εφαρμόζονται στο σύνολο των αγαθών που έχει κανείς στην κατοχή του ε, στην Ένωση όπου και αν βρίσκονται αυτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί δίνεται έτσι μια άθεση στην ανάπτυξη των οικογενειακών θεμάτων. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται ο κατάλογος των ομιλητών και καλό τον Επίτροπο να, βράσει, να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μετά από πολλά χρόνια περίπλοκων διαπραγματεύσεων, 18 χώρε μέλη εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στην ενισχυμένη συνεργασία. Ε, εγώ πιστεύω ότι και άλλε θα συμμετάσχουν. ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει με θετική ψήφο τους δύο κανονισμούς που διευκολύνουν τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών αποδομώντας νομικά εμπόδια. Είτε πρόκειται για έγκαμα ζευγάρια είτε πρόκειται για καταχωρισμένες σχέσεις θα τους επιτρέψει να ρυθμίζουν καλύτερα τις υποθέσεις τους. Ζητώ και από τις χώρες μέλη που δεν το έχουν πράξει ως τώρα να συμμετάσχουν στην ενισχυμένη συνεργασία διότι όσο περισσότερες χώρες μέλη συμμετάσχουν, τόσο περισσότερα εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών θα ωφεληθούν από τις ρυθμίσεις αυτές. Τέλος, ο κύριος Καβαντά λαμβάνει τελευταίος τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για απόψε θα είναι τα τελευταία λόγια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσία το Συμβούλιο, τις υπηρεσίες του, τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έθεσαν τέρμα σε έξι χρόνια ανισοτήτων. Γιατί το λέω αυτό, γιατί χρησιμοποιώ τον όρο ανισότητα. Διότι 18 χώρες μέλη δέχθηκαν να συνάψουν ας πούμε ένα σύμφωνο, πάντως να υπογράψουν τον ίδιο κανονισμό για τα έγκαμα ζευγάρια και τα καταχωρισμένα ζευγάρια, είτε πρόκειται για άντρα γυναίκα, είτε πρόκειται για ομοφυλόφιλα ζευγάρια, το έπραξαν αυτό διότι διεπίστωσαν ότι στις χώρες τους υπάρχει μια σχετική ανάγκη, μια ζήτηση. Δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν εκτός νόμου και σε σύγκρουση με διεθνή συστήματα όπου κανένας άνθρωπος μόνος του ακόμα και αν έχει ένα καλό συνήγορο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις περιπλοκότητες που προκαλούν τόση δυστυχία. Και μιλώ για 16 εκατομμύρια ζευγάρια, 32 εκατομμύρια ανθρώπους είτε είναι ε, παντρεμένοι είτε είναι σε καταχωρισμένες σχέσεις. Και επομένως 64 εκατομμύρια αν βάλετε και τους ε, ε, γονείς τους. Πρόκειται για πραγματικά καυκική υπόθεση. Ε, είμαι λοιπόν ιδιαίτερα ευγνώμων για την πολιτική βούληση που έδειξαν τα δύο ε, άλλα ε, συναρμόδια θεσμικά όργανα. Οι ε, μου και εγώ είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Γιατί καθυστέρησαν τόσο πολύ οι διαπραγματεύσεις αυτές, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τάχθηκε περισσότερο υπέρ της ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων, των αγαθών και των υπηρεσιών και λιγότερο των υποθέσεων των ζευγαριών. Καθυστερήσαμε λοιπόν πολύ. Τελικώς ξεπεράσαμε τα εμπόδια και καταλήξαμε τη συμφωνία αυτή. Έχω να πω δύο μικρά πράγματα ακόμα. Πρώτο, το κείμενο αυτό αμφισβητεί την επικουρικότητα, όχι, ουδόλως. Αντι, αντιθέτως, όσοι δεν επιθυμούν να δεν συμμετέχουν σε αυτή την ενισχυμένη συνεργασία των 18. Και όσοι έχουν πολίτες στην επικράτειά τους, όσες χώρες έχουν πολίτες στις επικράτειές τους, που ωστόσο ζουν σε άλλη χώρα που δεν επιθυμεί να τροποποιήσει το οικογενειακό δίκαιο, θα μπορούν να την χάνουν προστασία σε εφόσον απευθυνθούν σε δικαστήριο άλλη χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι καταλήξαμε σε ένα κείμενο το οποίο στην πραγματικότητα έχει ε, μια, ε, διέπεται από μια απλότητα και στην ουσία διακόπτει η πρόεδρος με το σφυράκι της. Τελειώνω κυρία Πρόεδρε. Θα έχουν τη δυνατότητα λοιπόν οι πολίτες να δουν εάν όντως τους ωφελεί η ρύθμιση αυτή και τότε να εξυπηρετηθούν από αυτήν, αλλιώς να την αρνηθούν. Ευχαριστώ όλες και όλους. Εδώ λίγη λέει η Πρόεδρος η κοινή συζήτηση και θα ψηφιστεί το κείμενο